Do la parola al collega. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Μύροσλαβ Μικολάτσης για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a dostupnej literatúry Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λόγω του όταν έγιναν 48 με 89 κομμουνιστικό καθεστώ στη Σλοβακία καταδίκαση 71.000 ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος για να ε, θυμηθούμε τους ανθρώπους αυτούς παρά μόνο με την διεύρυνση του χώρου δικαιοσύνης και ελευθερίας εκεί που θεωρείται πολυτέλεια αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε μέχρι στιγμής Ανησυχώ για την κατάσταση των πολιτικών κρατούμενων στην Κούβα και γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα να, να αναλάβουν όλα τα μέτρα για να απελευθερώσουν τους ανθρώπους αυτούς. Ε... Πρόεδρος Διακόπτη, παρακαλώ να βγείτε ήσυχα για να μπορούν οι συνάδελφοι να μιλήσουν. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Φίλι Κάτσμαρεκ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι, εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος στην για την Κούβα και δεν καταλαβαίνω γιατί οι φίλοι του Φιδέλ Κάστρο υποστηρίζουν αυτή τη χρεοκοπημένη ιδέα της επανάστασης. Χρειάζονται και άλλα θύματα του καθεστώτος για να μάθουν όλοι ότι χρειάζεται αλλαγή στην Κούβα. Καμιά φορά τα θύματα συμβάλλουν στην ιστορική αλλαγή. Το ίδιο θα γίνει και εδώ φαίνεται. Ελπίζω να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα όμως του καθεστώτος που θα οφείλονται στην ανικανότητά του να αλλάξει δεν δέχομαι το γεγονός ότι πολλοί υποστηρίζουν το καθεστώς αυτό νομίζω ότι είναι λάθος και λάθος αλληλεγγύη δεικνύουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε τι πέτυχε η Κούβα αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε και τις ελλείψεις της ο κύριος Μαρία Μόνης Ντεουρκουίτζα η κυρία Μαρία Μουνίθ Τεουρκούιθα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της κυρίας Μουνίθ για να εξηγήσω ότι η ψήφος της ε, Ισπανικής Αντιπροσωπείας στην τροπολογία υπαριθμών 2 της ε, Ενωτικής Αριστεράς ήθελε να απορρίψει αυτή την ε, τροπολογία, διότι παρά το γεγονός ότι ζητούσε υποστήριξη από την Ισπανική Προεδρία για τα θέματα της Κούβας, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να προσυπογράψουμε την τροπολογία μιας ομάδας η οποία διαχώρισε τη θέση της από το ψήφισμα. Εμείς λοιπόν, επειδή προσυπογράψαμε το ψήφισμα, δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε μία μερική τροπολογία στο ίδιο ψήφισμα. Και επίσης γιατί η τροπολογία υπαριθμών 2 της Ενωτική Αριστεράς δεν ανταποκρίνεται στη θέση της Ισπανικής Προεδρίας, η οποία αναζητεί συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναθεωρήσει το πλαίσιο των σχέσεων με την Κούβα, αλλά δεν θέλει απόλυτη ρήξη της, ε, των σχέσεων, όπως λέει αυτή η τροπολογία κατά γράμμα. Γι' αυτό απορρίψαμε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουζάννα Ρόιτοβα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ήταν τιμή για μένα να μπορέσω να υποστηρίξω το ψήφισμα για τους κρατούμενους στην Κούβα. Όχι μόνο γιατί εγώ προέρχομαι από μια τέλος κομμουνιστική χώρα, αλλά και λόγω μιας συνάντησης που είχα με τους αντιφρονούντε στην Κούβα όπου ενημερώθηκα παραδείγματος την κατάσταση του γιατρού Φεραίρα και παρουσίασα επίσης ε, το, στο κοινοβούλιο την φοβερή κατάσταση του συστήματος δημοσίας υγείας. Αν δεν έχει κανένα δολάρια δεν παίρνει καθόλου φάρμακα. Ο Σφερέρα βοήθησε τους ανεφερονούς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τώρα συνελήφθηκε ο ίδιος. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή το ψήφισμα που είναι τόσο έντονο ενεκρίθη και καλεί όλους να τηρήσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων εκεί στην Κούβα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λανάν, για ένα λεπτό πάντα. Πρόεδρε, πριν από 30 χρόνια, όταν ακούγαμε να πέφτουν τα τύχη και να βλέπουμε σήμερα ακόμα όμως ότι ο, ο, ο κύριος Κάστρο εξακολουθεί να είναι ηγέτης της Κούβα το κομμουνιστικό καθεστώς ε, που είναι εκεί κρατιέται από τον, ε, την, το αμερικανικό μπλοκό που τους επιτρέπει να κατηγορήσουν τους Αμερικανούς για τα οικονομικά τους ε, προβλήματα και επίσης η ενοχή ορισμένα στην Ευρώπη και ορισμένα εδώ μέσα στο, σώμα που έχουν φρικτά διπλά στάνταρτ και λένε ότι είναι καλή η Κούβα γιατί παράγει ε, μπαλαρίνες και γιατρούς. Έχει περάσει η εποχή των t με τον εβάρα Θα πρέπει να έχουμε μια πιο υποδομητική και σωστή στάση. Ο κύριος Φίλιπ Κλάις τώρα. Για ένα λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Είναι επικριτικό του καθεστώτος της Αβάνας, αλλά θα ήθελα να τονίσω με την ευκαιρία αυτή ότι θέλω να καλέσω το Συμβούλιο να, να σταματήσει, να πάψει αυτή την πρωτοβουλία του ε, των σχέσεων με την Κούβα γιατί πρόκειται για μια κομμουνιστική δικατατορία και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Καλό λοιπόν τους εκπροσώπους του να μην συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές ομαλοποίησης όπως έκανε τελευταία η Κομισιόν όπου ο Επίτροπος Μισελ είχε πάει στην Κούβα και δεν ε, εξέφρασε καμία επίκριση για την έλλειψη δημοκρατίας. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο για την Ένωση να δημιουργεί αδελφικές σχέσεις με κομμουνιστικά καθεστώτα. Ο κύριος Τσάνεσκι. Είναι παρόν. Παρόν. Όχι. Ε, τότε δεν υπάρχουν άλλες ευεξηγήσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι στη σε διάταξη. Να περάσουμε τώρα στο θέμα των τεχνολογιών ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακα να δώσω το λόγο στον κύριο Καλινόφσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αλλά θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών η χρηματοδότηση της προσπάθειας αυτής πρέπει να γίνει και από ιδιωτικούς όρους. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Ευρώπης το δικαιώνει αυτό. Οι κλιματικές αλλαγές και η σπάνης των ενεργειακών πόρων δικαιολογούν απόλυτα τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Είναι και μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, για την Ήπεθρο, ιδιαίτερα ως προς την ανάπτυξη ανανεωσίμων πηγών. Η Μπρεζίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ε, επενδύσεις υπέρ των τεχνολογιών ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εγώ υπερψήφισα γιατί θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει σε μια καινοτομική οικονομία που θα έχει πολύ συγκεκριμένους και καλούς στόχους και ελπίζω ότι η Κομισιόν μέχρι το 2011 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορέσει να ε, υποβάλει προτάσεις για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη εφιών δικτύων. Θα μπορέσουμε έτσι νομίζω να ε, ενισχύσουμε και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την ενίσχυση της ε, οικονομίας, με τη χορήγηση συμπληρωματικών δανείων στον τομέα αυτό και διεύρυνση των εγγύσεων για τα δάνεια. Αρνούμε το θέμα της τεχνολογίας με χαμηλότερη ε, εκπομπή ε, άνθρακος να χρησιμοποιηθεί για μια επίθεση κατά της ελληνικής ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Μαρκ Κρομπάντ. Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, nie mogłem poprzeć tej rezolucji, chociaż ona... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν ξεφράστην υπέρ του ψηφίσματος αυτού αν και το θέμα είναι ουσιώδες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά το ψήφισμα ε, προβλέπει υπερβολική χρηματοδότηση επιλεκτικά για πράσινους ενεργειακούς τομείς. Πράσινους. Και δεν έχει επιδειχθεί απαραίτητη ενεργειακή αλληλεγγύη με χώρες που βασίζουν την ενέργειά τους στον άνθρακα όπως η Παλανία Νομίζω ότι για να υπάρξει μία πιο μαλακή μετάβαση προς την πράσινη οικονομία δεν πρέπει τόσο απότομα μέτρα να λάβουμε γιατί δεν μπορούμε να καταργήσουμε την ε, τεχνολογία του άνθρακα από τη μια μέρα στην άλλη. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σοφία Αλκόνιο. Όχι, ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ξύνθια έπληξε βία τη Γαλλία. Περίπου 60 άνθρωποι πέθαναν και εκατοντάδες χιλιάδων υπέστησαν σημαντικές ζημίες. Μπροστά σε αυτό το δράμα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φανεί υποδειγματική και γι' αυτόν τον λόγο προσωπικά ενεπλάκην στη σύνταξη του ψηφίσματος που ζητάει από την Ευρωπαϊκή ε- να είναι πιο δραστήρια. Σημαντική δηλαδή οικονομική βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης. Εάν με βάση το δράμα αυτό η περιοχή που ατού Σαράντ Σαράντ Μαριτίμ, Πέιντε Λαλουάρ και Βρετάνη ζητήσουν αλλαγή του προγραμματισμού των δαπανών τους σε συγχρηματοδότηση με το Φεντέρι το FSU τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε τις, τα αιτήματα αυτά να τα μελετήσει με πολύ μεγάλη προσοχή και να τα με θετική αντιμετώπιση. Αλλά και πέρα από το ψήφισμα, γιατί όπως και οι άλλοι συνάδελφοι της προεδρικής πλειοψηφίας, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματική, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σώμα πολιτικής ε, που θα ήταν πολύ σημαντική βοήθεια για την αντιμετώπιση τέτοιων θεών κύριος Κέλλη είχε ζητήσει να μιλήσει για, την προηγούμενη, για το προηγούμενο ψήφισμα ε, όλος εξαιρετικός θα το δεχτούμε αλλά την άλλη φορά όχι δεν, δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα Ευχαριστώ πρόεδρε σύντομα θα ήθελα να πω ότι καιρό είναι πια να υπάρξει ένα τελειωτικό έγγραφο νομοσχέδιο για τα ενεργειακά προβλήματα τι θέλουμε να κάνουμε για το μέλλον, δηλαδή πώς θα μεταφραστούν οι αναλύσεις μας σε συγκεκριμένη έρευνα. Γιατί έχουν ακουστεί πολλές αμφιβολίες και σκεπτικισμός. Και δεν έχουν λυθεί όλα αυτά από την σημερινή συζήτηση. Σε αυτή τη διακοσιωστή απέτειο της ανεξαρτησίας της Λιθουανίας και της Εσθονίας πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Ε? Ωραία, θα συνεχίσουμε στις 3. Διακόπτω τη συνεδρίαση. Grazie, ε,